Εγκρίνεται η συμβαστική 1. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 203 του κυρίου Νταντά. Ποιο είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 204 υπέρ. Εγκρίνεται. 205 υπέρ. Εγκρίνεται. Ή μάλλον συγγνώμη, ε, κατά. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10 της ΔΕΒΕ. Ποιος είναι υπέρ της ΔΕΒΕ 10. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Πάμε στην ΕΒΗ 10. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικό έλεγχος για την τροπολογία 10 τη Επιτροπής Περιβάλλοντος. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλο ψηφοφορία και απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλο ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. εγκρίνεται. Και πάμε στη συμβαστική τροπολογία 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 238. Ποιος είναι υπέρ? Εγκρίνεται. Μαζί με τη 239 που είναι πανομοιότυπη. Τροπολογία 240 και 241. Ποιος είναι υπέρ? Εγκρίνονται. Τροπολογίες 242 και 243 υπέρ. Εγκρίνονται. Τροπολογία 244 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία ονομαστικά για την τροπολογία 244. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12 της ΔΕΒΕ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 14 υπέρ. Εγκρίνεται. Πάμε στη 246 του κυρίου Μέλο. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 248 και 249 μαζί. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνονται. Πάμε στη συμβαστική τροπολογία 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Συμβαστική 7. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Πρέπει να περάσουμε κάνα δύο σελίδες. Άρχεται η ψηφοφορία για τη συμβαστική τροπολογία παριθμών 8. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική τροπολογία παριθμών 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. εγκρίνεται. Και πάμε στην 323 τροπολογία. Τροπολογία 323 του κυρίου Καπούτο. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 319. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και πάμε στην τροπολογία 20 του εισηγητού. Ποιος είναι υπέρ? Εγκρίνεται. Τροπολογία 341. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Απορρίπτεται μάλλον, αλλά στο ελέγξουμε καλού κακού. Άρχεται η ψηφοφορία για την 341. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ευτυχώς που το ελέγξαμε. Τροπολογία 21. Ποιος είναι υπέρ, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 339. Μαζί με την 340 που είναι ταυτόσιμες. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. Τροπολογία 11α. Συμβαστική. Άρχεται η ψηφοφορία. Συμβαστική 11α. Τέλος ψυχοφοριας Εγκρίνεται. Συμβαστική 12. Ή μάλλον 348. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 349 υπέρ εγκρίνεται. 350 τώρα. Ποιο είναι υπέρ της 350 τροπολογία Υπέρ εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική τροπολογία 12 τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία για τη συμβαστική 12. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 378 της κυρίας Αγγιλέρα. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 13. Ποιος είναι υπέρ. Συγγνώμη, θα χρειαστεί να επαναλάβουμε την ψηφοφορία για την τροπολογία για τη συμβαστική 12, γιατί χρειάζεται ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία, για τη συμβαστική τροπολογία 12, ονομαστική ψηφοφορία. Μα την κάναμε ήδη, λέει κάποιος από την αίθουσα. Ναι, ναι, το ξέρω ότι ψηφίσαμε. 16 υπέρ, 18 υπέρ, 16 κατά. Όχι, όχι, δεν είναι ε, για τη 12, λέω. Ονομαστική κλίση. Τέλος ψηφοφορίας. E, Συγγνώμη, υπήρξε ένα τεχνικό πρόβλημα. Τεχνικό λάθος δεν πάτησε τη σωστή, το στο κουμπί η γραμματεία ότι ήταν ονομαστική ψηφοφορία και έπρεπε να την επαναλάβουμε. Γι' αυτό και χρειάστηκε να επαναλάβω ως ονομαστική ψηφοφορία την ψηφοφορία για την συμβαστική τροπολογία 12. Γι' αυτό σας ζήτησα να επαναλάβουμε. Έπρεπε να ξαναψηφίσουμε ονομαστικά την 12. Υπερψηφίστηκε η 12. 3,78 τώρα. Okay. Okay, powtarzam, głosujemy poprawkę. Επαναλαμβάνω. Ψηφίζουμε με ονομαστική κλίση τη συμβαστική τροπολογία 12. Το είπα και πριν, δεν με καταλάβατε. Ονομαστική ψηφοφορία για τη συμβαστική 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην τροπολογία 378 Ψηφίζουμε την τροπολογία 378 της κυρίας Αγγιλέρα. Ποιος είναι υπέρ, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 407 του κυρίου, του κυρίου Νταντά. Ποιος είναι υπέρ? Ευχαριστώ, εγκρίνεται. 408. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 410 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 14α. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται και πάμε στη συμβαστική τροπολογία 15. Συμβαστική 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 419 τον Ανδρίο Γκλοανέκ και άλλων. Ποιος είναι υπέρ, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 16, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17, συμβαστική. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στο 474. 474. Μερικές σελίδες παρακάτω. Χαίρομαι που προχωράμε έτσι γρήγορα. 474 λοιπόν, τον Λουαζό και Κολομπιέ. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 475 υπέρ, εγκρίνεται. 476 υπέρ. Εγκρίνεται. 477 υπέρ. Εγκρίνεται. 478 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 18. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 19. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 20. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 21. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Συμβαστική τροπολογία 22. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 23. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 23 λέει ο πρόεδρος. Λάθος, λάθος λέει. Συγγνώμη, 24, 24. Την 23 την υπερψηφίσαμε. Άρχεται η ψηφοφορία για τη συμβαστική 24. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στη 532. Τροπολογία 532 του κυρίου Νταντά. Ποιος είναι υπέρ εγκρίνεται. 533 υπέρ, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 25, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 26, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 27. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 28. 28. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 29. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και πάμε στην τροπολογία 564. Αντριέ και άλλων. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 556 και 557. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνονται. 429 και αυτή ήταν μαζί με τις προηγούμενες δύο. Συμβαστική τροπολογία 30 τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 31. Άρχεται η ψηφοφορία για την 31 συμβαστική. Τέλος. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 57 τώρα του εισηγητού. Ποιο είναι υπέρ, εγκρίνεται. 58 υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικό έλεγχος για την τροπολογία 58, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. Τροπολογία 59. Ποιο είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Κατά. Υπέρ. <laughs> Εγκρίνεται. 567 υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 60 του εισηγητού υπέρ. Εγκρίνεται. 61 του εισηγητού. Εγκρίνεται. 568. Ποιος είναι υπέρ? Εγκρίνεται. 569. Μαζί με την εβ 3 υπέρ. Εγκρίνονται. 571 και 572. Ποιος είναι υπέρ? Κατά ηλεκτρονικό έλεγχο Άρχεται η ψηφοφορία για τις τροπολογίες 571 και 572. Τέλος ψηφοφορία. Εγκρίνονται. Τροπολογίες 573, 574 και 575. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. 576 και 577. Ποιος είναι υπέρ. Κατά απορρίπτονται. 578. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 578. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Δεύε 13. Ποιος είναι υπέρ κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 32. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 581. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ονομαστικά. Για το 581. Τέλος. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 33. Άρχεται η ψηφοφορία. Otwieram głosowanie. Kompromis 33. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 33α νέα. Άρχεται η ψηφοφορία για την 33α νέα. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 34. 34. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 35. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 36. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 37. Συμβαστική τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 38. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 39. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και πάμε στην τροπολογία 68 του εισηγητού. Ποιος είναι υπέρ? Εγκρίνεται. 69 του εισηγητού και πάλι υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 40. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 41. 41. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και πάμε στη συμβαστική τροπολογία 42. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 43. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και αυτή και περνάμε στην τροπολογία 693 υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 44. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 45 συμβαστική. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και πάμε στη συμβαστική τροπολογία 46. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 720 του κυρίου Νταντά. Ποιος είναι υπέρ? Εγκρίνεται. 721 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 721. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. 722. Ποιος είναι υπέρ, 722. Εγκρίνεται. 723. Ποιος είναι υπέρ, εγκρίνεται. 724 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 724. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 47. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 48. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 49. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 50. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 51 συμβαστική τροπολογία. Ποιος είναι, ε, άρχεται η ψηφοφορία, συγγνώμη. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 52. άρχιτε ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 53. άρχιτε ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 54. άρχιτε ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Η 754 καταπίπτει. Πάμε στην συμβαστική 55, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 56. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 762. Ποιος είναι υπέρ? Εγκρίνεται. 57 συμβαστική τροπολογία, άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην τροπολογία 19 της Επιτροπής Ρέτζι. Ποιος είναι υπέρ, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 58, άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 781, 783, 107, 782 και MV50. Ποιος είναι υπέρ? Εγκρίνονται. 59. Ποιος είναι υπέρ? Ε, μάλλον συμβαστική τροπολογία. 59. Αρχιτή ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται η συμβαστική τροπολογία και πάμε στη συμβαστική τροπολογία 60. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται η συμβαστική τροπολογία 60. Τώρα, συμβαστική τροπολογία για τις αιτιολογικές σκέψεις. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και πάμε στην τροπολογία 110 στη σελίδα 116. 110 τροπολογία. Λίγες σελίδες παρακάτω μαζί με την κοντ 1. Τροπολογία 110 και τροπολογία 1 της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνονται. Τροπολογία DV2. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 114 τώρα. Και κοντ 2. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνονται. Ρέτζι 4. Ρέτζι 4. Ποιος είναι υπέρ? Ρέτζι 4. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 4 της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Όλα καλά, όλα καλά. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 4 της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ρέτζι 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Ρέτζι 4. Μια στιγμή Άλλο γράφει, άλλο ψηφίζει. Ο κύριος Νταντέν, ας το ελέγξουμε. Ρέτζι 4. Ψηφίζουμε τη Ρέτζι 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 118. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 125 ή όχι. Όχι, όχι. ΔΕΒΕ 6 πρώτα. Τροπολογία 6 της Επιτροπής Ανάπτυξης. ΔΕΒΕ 6. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Μια στιγμή να συνεννοηθούμε. Εκατόν τριάντα έξι του κυρίου Μπούντα. 136. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 147. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 7. ποιο είναι υπέρ. Εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 8. ποιο είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Εκατόν εβδομήντα Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 182. έμβιο 8 και ντεβε 7 λέει ο πρόεδρος. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τις τρεις τροπολογίες, άρχιτη ψηφοφορία. Do you mind repeating? Πρόεδρε, ε, έχετε την καλοσύνη να μας εξηγήσετε τι ακριβώς ψηφίζουμε. Τέλος ψηφοφορίας. Ο κύριος Άγνιου. Ψηφίσαμε τις τροπολογίες την τροπολογία 179 λέει ο πρόεδρος. Ε, sorry, sorry. Λάθος, λάθος, διορθώνει ο πρόεδρος. Λάθος, μια στιγμή, άργα, σιγά σιγά. Ψηφίζουμε τις τροπολογίες 182, MV8 και DV9. Εντάξει. Πάμε τώρα στην 187 υπέρ. Απορρίπτεται. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε που παρατείνω την διαδικασία. Σας ρώτησα τι ψηφίζουμε. Είπατε 182 και 187 αμέσως μετά. Ε, ποιο από τα δύο τελικά. Ψηφίσαμε τις τροπολογίες 182, mv 8 και DV9 με ηλεκτρονικό έλεγχο. Και τώρα θα ψηφίσουμε την 187 187. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Η γραμματεία δεν πρόλαβε να σημειώσει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας των τριών τροπολογιών 182, MV8 και DV9. Οπότε θα επαναλάβουμε την ψηφοφορία. Πού είναι το πρόβλημα? δεν πρόλαβε η γραμματεία να σημειώσει το αποτέλεσμα τη ψηφοφορία των τριών τροπολογιών, 182, MV8 και DV9. Ξαναψηφίζουμε λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλο ψηφοφορία. Απορρίπτονται. Τροπολογία 187 ψηφίσαμε. 191 του κυρίου Νέκοφ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Μάλλον ηλεκτρονικός έλεγχος για την 191. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Αυτή ήταν η τελευταία τροπολογία. Και ψηφίζουμε το σύνολο της έκθεσης. όπως έχει τροποποιηθεί, με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ονομαστική ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Σιγητά. Κύριε Αντρέα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που ετοίμασαν την ψηφοφορία. Όπως είπα και στην αρχή, αν αυτή η ψηφοφορία καθορίζει και τις επόμενες, είναι καλός ιονός για το μέλλον της μεταρρύθμισης. Δεν θα πω τα ίδια. Θέλω να ευχαριστήσω όλους και όλες για την εντατική προσπάθεια που καταβάλαμε αυτούς τους μήνες. Ευχαριστώ λοιπόν την εφή ψηφοφορία που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια αυτή. ΚΟΑ για την επόμενη θητεία. Αφήνουμε αυτό το έργο στους διαδόχους μας, ούτω ώστε να καταλήξει σε αποτελέσματα αυτή η εργασία. Και ευχαριστώ όλους. Proszę przyjąć, proszę przyjąć w nas μπορείτε να δεχτείτε τις ευχαριστίες όλων μας, κύριε Σιγητά, και συγχαρητήρια και ευχαριστίες για τους και οδησηγητές, τους σας, την γραμματεία, όλους όσους συνέβαλαν στην εκπόνηση αυτής της έκθεσης. Νομίζω ότι είναι αξιόλογο αυτό το έγγραφο, αξιόλογη έκθεση. Σας ευχαριστούμε θερμά, οπότε μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Ξαναευχαριστώντας σας και πάλι. Μας έμεινε και χρόνο συνεδρίες, οπότε αν θέλει κανείς το λόγο, πολύ ευχαρίστω. Δεν βλέπω κανένα να θέλει το λόγο. Σας εύχομαι καλό βράδυ και ραντεβού αύριο στις 9 το πρωί. Α, 9 πρέπει να βγάλουμε αναμνηστική φωτογραφία. Ευχαριστώ και πάλι και τη γραμματεία. Σας ευχαριστώ όλους θερμά. Νομίζω ότι πήγαν όλα καλά. Οπότε βάζουμε πλώρη για τις επόμενες εκθέσεις. Ελπίζω αύριο να μην ε, χαλάσει η κάρτα ψηφοφορίας της κυρίας Εράς Γκαρσία, γιατί σήμερα της έσπασε η κάρτα. Σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.